Συνάδελφοι, ας περάσουμε στο επόμενο θέμα της μερίσιας διάταξης, το πρωτόκολλο της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιορδανίας σε σχέση με τις γενικές αρχές που διέπουν συμμετοχή της Ιορδανίας στο πρόγραμμα της Ένωσης. Θα μιλήσουμε για τις τροπολογίες, για την ε, συμμετοχή, του Χασιμητικού Βασιλείου της Ιορδανίας για τη συμμετοχή στα προγράμματα της ε, Ένωσης. Επτά τροπολογίες έχουν ε, υποβληθεί. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Νέιτς για να μας ε, μιλήσει για τις τροπολογίες αυτές. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ για την ε, εισαγωγή αυτή. Δεν χρειάζεται να δαπανίσουμε και πολύ χρόνο για να αποφασίσουμε. Νομίζω ότι τα στοιχεία αυτά είναι ε, σαφή. Εάν λοιπόν συνενέσει το Κοινοβούλιο, για το πρωτόκολλο αυτό, το προσχέδιο πρωτοκόλλου σημαίνει ότι η Ορδανία θα έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών και σε αυτή την περίπτωση θα αποστείλουμε ένα σαφές ε, μήνυμα στο βασίλειο της Ιορδανίας ότι δηλαδή προτιθέμεθα να υποστηρίξουμε την ε, Ιορδανία μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης αλληλεγγύης και αυτό τη στιγμή που η Ορδανία αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες λόγω των προβλημάτων της ε, περιοχής. Επτά τροπολογίες έχουν ε, υποβληθεί, κύριε Πρόεδρε, όπως προαναφέρατε. Σύσταση προς τους συναδέλφους είναι να δεχτούμε όλες τις τροπολογίες εκτός από την 4 και 5 και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που υπέβαλαν τις ε, τροπολογίες και έτσι συνεισέφεραν για τη βελτίωση της έκθεσής μου αυτής. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Νέιτς. Συνάδελφοι, υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να λάβει το λόγο. Ο κύριος Σαλαφράγκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εντάχει απλώς να συγχαρώ την κυρία Νέιτσε και να πω ότι η κυρία Σάιφη είναι η δική μας ε, σκιώδης που δεν παρίσταται εδώ γιατί βρίσκεται σε άλλη συνεδρίαση και εξ ονόματός της θα ήθελα να πω ότι από πλευρά της δικής μας ε, πολιτικής ομάδας δεν έχουμε πρόβλημα να αποδεχτούμε αυτή την έκθεση. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες ως προς τις τροπολογίες, αλλά εν πάση περιπτώσει θα υπερψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Ευχαριστούμε κυρία Σαλαφράνκα. Από τους σοσιαλιστές θα ήθελε κάποιος να λάβει το λόγο ή από τους φιλελευθέρους, από άλλες ομάδες. Δεν βλέπω να ισχύει κάτι τέτοιο. Μπορούμε λοιπόν... Κυρία Νέιτς, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Όχι, λέει η κυρία Νέιτς, φαντάζομαι ότι αύριο θα γίνει η ψηφοφορία και σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας. Ευχαριστώ πολύ, διακόπτουμε και μετά θα ασχοληθούμε με τις υποψηφιότητες για το βραβείο Ζαχάροφ. Ευχαριστώ.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

Mrs. Nielsen is not here. The Greens, please. I have here Mrs. Nielsen, but is not here. Oui, je remplace Madame Kiel Nielsen qui doit arriver mais qui a eu un problème de train. Donc je la remplace au pied levé.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 very much, Mr. Marek Migalski, for the nomination of Ales Bialatsky, Eduard Lobau, and Mikola Statkevich on behalf of all Belarusian political prisoners. This nomination was supported also by Filip Kaczmarek, Mr. Protasevich, and 39 other members. Mr. Migalski, please. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście ta nominacja została poparta przez